As you know, our colleague Mr. Danjan left today Libya with an ad hoc mission. Ο κ. Ντανζάν πήγε στη Λιβύη με την Επιτροπή Ad hoc. Και γι' αυτό θα προεδρεύσω σήμερα. Βλέπετε ποιες είναι οι γλώσσες Σας θυμίζω ότι η προτεραιότητα στη χρήση των γλωσσών έχουν τα τακτικά μέλη. Και ταυτόχρονα σας θυμίζω ότι αναμεταδίδεται η συνεδρίαση στο διαδίκτυο. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρείται δεκτή η σε διάταξη. Αν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σχετικά με τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων, θεωρούνται δεκτά. Δεν έχω καμία ανακοίνωση από πλευράς Προεδρείου και θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Eurojust Lex. Να καλωσορίσω τον κύριο Χαμπέρ, ο οποίος είναι διοικητής στα πλαίσια της CPCC και τον κύριο Λάτσλο Χούσακ που είναι ο υπεύθυνος της αποστολής Eurojust Lex στο Ιράκ. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της διαχείρισης κρίσεων και στα πλαίσια της ΚΕΠΑ έχει ξεκινήσει να ασχολείται με την αποστολή αυτή αποφασίστηκε να παραταθεί η ισχύ της μέχρι τις 30 Ιουνίου. Πέρυσι διορίστηκε ο στρατηγός Χούζεκ, αρχηγός της αποστολής επιτόπου στο Ιράκ. Το 2003 ξεκίνησε η δεύτερη, ο δεύτερος πόλεμος του Ιράκ, Το Δεκέμβριο του 2011 οι τελευταίοι ξένοι στρατιωτικοί σχηματισμοί εγκατέλειψαν τη χώρα. Οι εσωτερικές δυνάμεις ασφαλείας ελέγχουν κατά το μάλλον ή τον την κατάσταση στην χώρα. Και αυτός είναι ο λόγος στα πλαίσια των οποίων στα πλαίσια των συνθήκων αυτών μάλλον καλείται και η, Euro, ε, και Eurojust Lex να φέρει πέρα στην αποστολή της. Υπάρχουν τα θέματα αντιπαραθέσεων μεταξύ Σία και Σούνη, υπάρχει το θέμα της κουρδικής α, ε, ε, περιοχής που κατοικείται κυρίως από Κούρδους. Γενικά οι επαφές ανάμεσα στις κοινότητες της χώρας μπορεί να αποβούν ιδιαίτερα τεταμένες ορισμένες φορές και γι' αυτό και η αποστολή Eurojust Lex είναι πολύ δύσκολη. Mark, allow me και μετά από αυτές ε, τις ε, παρατηρήσεις τις εισαγωγικές θα δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους. Δίνουμε προτεραιότητα σε αυτούς οι οποίοι δουλεύουν επιτόπου στις αποστολές και γι' αυτό στρατηγοί δεν σας δίνουμε το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε κύριοι βουλευτές, αγαπητοί φίλοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, διότι είναι η πρώτη φορά που απευθύνομαι στην Επιτροπή σας. Τέσσερις μήνες μόλις ε, ανέλαβα τα καθήκοντα του επικεφαλής της αποστολής EU Just Lex στο Ιράκ. Πρέπει να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη κάπη της Ιράκινης ιστορίας μετά την απόσυρση των ε, στρατευμάτων ε, τον ΙΠΑ το προηγούμενο Δεκέμβριο από το Ιράκ πλέον ε, παίρνει τα ενία της χώρας του ο λαός του Ιράκ και επιτυχία, επιθυμία της μεγάλης πλειοψηφίας είναι να προοδεύσει η χώρα προς ένα δημοκρατικό καθεστώς που θα αγγιάται τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους. Θα συμφωνείτε φαντάζομαι ότι και η Ευρώπη θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτή την ιστορική προσπάθεια. Το EU Just Lex του Ιράκ είναι μία από τις πιο απτές ε, συνεισφορές ε, στις δημοκρατικές φιλοδοξίες του Ιρακινού λαού με την πολύτιμη συνεργασία υποστήριξη της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Ιράκ. Με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουμε να συνεργαστούμε για να προωθήσουμε την γενική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε την στήριξη των ε, μελών ε, ε, που συμμετέχουν στο θέατρο επιχείρηση αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε για να πετύχουμε τους στόχους μας στο ίδιο πλευρό με τους Ιρακινούς. Και θέλω να σας πω με χαρά ότι με καλωσόρισαν θερμά οι Ιρακινοί ομόλογοι μας σε όλα τα επίπεδα στις τρεις τοποθεσίες που είμαστε παρόντες, δηλαδή στην πρωτεύουσα την Βαγδάτε, την Ερμπίλ ε, που είναι η κουρδική περιοχή και στην Πάσραφ στο Νότο. Όπως γνωρίζετε, όταν ξεκίνησε τις εργασίες της το 2005 η αποστολή, η κατάσταση ασφαλείας δεν επέτρεπε την άμεση ανάπτυξη στο θέατρο επιχειρήσεων και γι' αυτό έπρεπε κυρίως να δραστηριοποιηθούμε σε άλλα ε, μέλη πολύ λίγη, πολύ μικρή χρονικά ήταν η παρουσία μας ε, στην ε, Βαγδάτη και μόνο το 2010 καταφέραμε να ε, διευρύνουμε την παρουσία μας και στην Ερμπίλ και στην Πάστρα δηλαδή. Η... Τα αρχηγεία μας μετέφεραν, με, τα μετεφέραμε στην Βαγδάτη το Φεβρουάριο του 2011. Έγινε η πρώτη ανάπτυξη και η υπόλοιπα αρχηγεία στρατηγική σταδιακά μεταφέρθηκαν. Το τέλος του Ραμαζανίου τον Αύγουστο του 2011 είχαμε πλέον τον μεγάλο όγκο των επιρρογνωμόνων μας ε, επιτόπου στη χώρα μέσα. Η διαδικασία αυτή ε, ήταν γεμάτη από προκλήσεις, αλλά πλέον ε, είμαστε επιχειρησιακοί, λειτουργούμε καλά, συνεργαζόμαστε όσο καλύτερα μπορούμε με τους Ιρακινούς και έχουμε συνεργασία και με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα σοφρανιστικά ιδρύματα. Έχουμε μια σταθερή παρουσία, 31 άνδρες και γυναίκες έχουμε και άλλοι 14 είναι στην Ερμπίλ και 9 στην Μπάσρα, όπου έχουμε εμείς εκεί 6 συναντέλφου. Η ανάπτυξη τη αποστολή μα στο Ιράκ κατάφερε με πολύ μεγάλη επιτυχία να δημιουργήσει καλές σχέσεις με τους τοπικούς ομολόγους η αποστολή αυτή, η You Just Lex, θεωρείται ναι με μία μικρή σε σύνθεση, αλλά ευέλικτη αποτελεσματική αποστολή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία για την αποστολή μας σε συνεργασία με τις Ερακινές Αρχές. Διοικητεύονται πολύ σημαντικά θέματα στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ άλλων, αλλά και πρόσβαση στη διπλωματικό καθεστώς, ελευθερία ε, κυκλοφορίας, μειωμένη έκθεση σε διάφορους κινδύνους. Είναι κάποιε από τι προκλήσει. Καταφέραμε να διαπραγματευτούμε ένα πολύ ικανοποιητικό σχέδιο συμφωνία που θα εξασφαλίσει στο προσωπικό μα και στι επιχειρήσει μα στο Ιράκ την απαιτούμενη προστασία. Η τελική συμφωνία αναμένεται σύντομα από την Ιρακινή κυβέρνηση. Αγαπητοί βουλευτέ υποτροπή, η EU Just Lex παρέχει και εκπαίδευση και ε, έλεγχο και συμβουλές. για να ε, αυτονομηθεί και το σύστημα ε, το δικαστικό στο Ιράκ. Έχουμε κάποιες δραστηριότητες ε, και σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η εκπαίδευση κατά κύριο λόγο πλέον μετά τη μεταφορά της αντιπροσωπείας μας στο Ιράκ γίνεται εκεί, επί τόπου. Για να σας δώσω λίγα παραδείγματα αστυνομική εκπαίδευση, για την τακτική έρευνα. Μεταξύ άλλων, και θέλουμε να βασιζόμαστε κυρίως σε επιστημονικές συμβουλές για την ε, ποινική έρευνα και ανάκριση και όχι σε προφορικές ε, καταθέσεις. Για τη σωματεμπορία τώρα. Οι ομόλογοι μας πλέον να παίρνουν τα ενία για να εντοπίζουν διάφορες μορφές εγκληματικότητας με τις οποίες δεν είναι ακόμη εντελώς εξοικειωμένοι. Για τη σοφρονιστική εκπαίδευση, στόχος μας είναι η αποκατάσταση των κρατουμένων, η βελτίωση των συνθήκων στις φυλακές, ώστε να πλησιάσουν τα πρότυπα τα δικά μας. Τις τελευταίες έξι μήνες διενεργήσαμε 34 εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε 455 αξιωματούχους 5.000 είχαν ήδη εκπαιδευτεί στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ε, στην ίδια τη χώρα, ε, σε συνάρτηση με τις ανάγκες της χώρας. Βέβαια, ε, πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν τεράστιες προσπάθειες και έχουμε και κάποιες ιστορίες επιτυχίας. Καταφέραμε να συνδυάσουμε ε, τις αστυνομικές δραστηριότητες με τις δραστηριότητες. Έχουμε μεγαλύτερη γυναικεία παρουσία και οργανώνουμε και την πρώτη δικαστική δραστηριότητα στο σχετικό ίδρυμα στη Βαγδάτη. Αυτά είναι μερικά από τα παραδείγματα της επιτυχίας που έχουμε να επιδείξουμε. Τους τελευταίους μήνες, αφού εξοικειωθήκαμε πλήρως με τις δυσκολίες που έχει το επιχειρή στο Ιράκ, μπορώ να σας πω ότι αξίζει ευχαριστειών η αντιπροσωπεία μας, η αποστολή, η You Just Lex, και ε, το έργο που έχετε επιτελεστεί και αυτό που θα επιτελεστεί θα μπορούσε να ε, πραγματοποιηθεί αν δεν είχαν κάνει τις προσπάθειές τους, γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση ασφάλειας. Φαντάζομαι, θα καταλάβετε και από το επαγγελματικό μου υπόβαθρο, ότι την εκπαίδευση τη θεωρώ κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ιδίως για τα θέματα ασφαλείας, ε, που είναι και η βασική μου αρμοδιότητα θα παρακολουθήσουμε πάρα πολύ προσεκτικά την κατάσταση για να δούμε μήπως επιδεινωθεί σημαντικά η κατάσταση με την απόσταση των Αμερικανικών στρατευμάτων. Ήδη έχουμε ξεκινήσει αυτόν τον έλεγχο και δεύτερον θα καταβάλουμε συνεχείς προσπάθειες ώστε να έχουμε ασφαλείς και κατάλληλες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις για τις δραστηριότητές μας. Αγαπητοί βουλευτές υποεπιτροπής, άμυνας και ασφάλειας. Η e Lex ε, στο Ιράκ ε, συνεργάζεται πάρα πολύ στενά ε, με τους ομολόγους μας από το Ιράκ, θέλω να, μάλλον από άλλες χώρες. Θα σας μιλήσω συγκεκριμένα για τη συνεργασία μας με τη ΣΥΠΑ. Δραστηριότητες κράτους δικαίου στο Ιράκ. Από το Υπουργείο Άμυναν πέρασαν στο Υπουργείο του Κράτους, στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά έχουμε στενή συνεργασία και με αυτό το Υπουργείο. Η Αμερικανοί ομόλογοι μας συμμετέχουν στο σχεδιασμό, ανταλλάσσουμε πληροφορίες, ε, διευκολύνσεις. Μαζί οργανώσαμε το φόρουμ ε, κράτους δικαίου στο Ιράκ. Γιατί καταλαβαίνουμε βέβαια ότι η βελτίωση κατάσταση στο Ιράκ ε, είναι προς αμοιβαίο όφελος και όχι μόνο, είναι μια επιτακτική επιχειρησιακή ανάγκη. Το ίδιο ισχύει βέβαια και με άλλους διεθνείς ομολόγους μας, με τους οποίους συνεργαζόμαστε στενότατα όπως είναι και η ευρύτερη οικογένεια του ΟΗΕ στο Ιράκ. Με χαρά μπορώ να σας ανακοινώσω ότι σύντομα η Νορβηγία θα είναι το πρώτο τρίτο κράτος το οποίο θα συνεισφέρει ε, στην αποστολή You Just Lex στο Ιράκ. Βέβαια, πριν να ολοκληρώσω, δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω ε, όλους σας που μου δώσετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω την ε, τρέχουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά την αποστολή αυτή που έχουμε στο Ιράκ. Αν με επιτρέπετε, Θα ήθελα να πω ότι η κοινή, ευρωπαϊκή, η κοινή ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας θα πρέπει να ανταποκρίνεται μεταξύ άλλων και στις ανησυχίες που εκφράζουν οι πολίτες της Ευρώπης. Θα ήθελα τώρα να ακούσω βέβαια τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας ερωτήσεις και με τα χαράς να απαντήσω σε απορίες σας. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you for... Ευχαριστώ για την ε, πολύ συνεκτική σας παρουσίαση και θα δώσω τον ε, λόγο εις ε, τον ε, κύριο Χάμπερ και στη συνέχεια θα υπάρξουν ερωταπαντήσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά σε αυτά τα οποία σας είπε ο επικεφαλής της αποστολής και θα σας πω ποια είναι η προοπτική των Βρυξελών διότι όπως ε, ήδη αναφέρθηκε ε, ε, ξεκίνησε η αποστολή και η κατάσταση συνέχεια χειροτέρευε. Εκείνη την εποχή ε, δεν μπορούσαμε να έχουμε μία αποστολή που να λειτουργήσει επί τόπου, αλλά δουλεύαμε από τις Βρυξέλλες ε, ε, καλώντας εδώ Ιρακινούς οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν όπως επίσης και από τα κράτη-μέλη τα οποία οργάνωναν εκπαιδευτικά προγράμματα. Και μετά μπορέσαμε να επανα τοποθετήσουμε την ε, αποστολή μας στο Ιράκ. Ο πρώτος ήταν ε, ε, αυτός ο, ο οποίος επανέφερε επί τόπου στο Ιράκ την αποστολή και προέβη στα μέτρα τα οποία ανέφερε ο Βρολαλίσας. Ε, βέβαια όλα αυτά ξεκίνησαν πριν από 7 χρόνια, αλλά ουσιαστικά είναι μια νέα μορφή και είναι νέα όσον αφορά τις ε, ε, τις προκλήσεις της διοικητικής Μέριμνας και όσον αφορά του Συρακινούς. Δηλαδή, ενώ τα κράτη-μέλη και, εσύ, και εσείς μπορεί να θεωρείτε ότι υπάρχει μία επιπλέον στρατηγική, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να σας προσφέρουμε, διότι εν πολλής πρόκειται για μία νέα αποστολή. Απ' την άλλη πλευρά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να γίνει αυτή η κίνηση διότι βελτιώθηκαν οι επαφές και η αξιοπιστία μας στους Ιρακινούς διότι είμαστε επιτόπου στην πράσινη ζώνη αλλά και εκτός της πράσινης ζώνης για εκπαιδευτικούς σκοπούς οπότε αναλαμβάνουμε τους ίδιους κινδύνους με αυτούς πράγμα το οποίο αυξάνει την αξιοπιστία της αποστολής μας. Σε σχέση λοιπόν με αυτή την κατάσταση πρέπει τώρα να υπάρξει ένας διάλογος με τις αρχές του Ιράκ και για μας τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας στρατηγικός διάλογος με το Ιράκ για να μπορούμε ε, να βρούμε ρεαλιστικούς στόχους γιατί ε, το Ιράκ είναι ε, μια τεράστια χώρα, δεν μπορούμε να την καλύψουμε ολόκληρη. Ξέρετε ποιες ήταν οι εξελίξεις μεταξύ το 2003-2004 όπου ένα μεγάλο μέρος των δυνάμεων ασφαλείας είχαν διαλυθεί και πρέπει τώρα να νοικοδομηθούν και να ανασυσταθούν. Οπότε είναι σαν ε, να προσπαθούμε να πετύχουμε έναν κινούμενο στόχο και ε, ε, πρέπει ανα πάσα στιγμή να επαναξιολογούμε πού πρέπει να επέμβουμε μέχρι ότου να μπορέσουμε να θεωρήσουμε ότι θα έχουμε ολοκληρώσει την αποστολή μας. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα από τις αποστολές στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν είναι ότι ο συντονισμός με τους άλλους παράγοντες που επεμβαίνουν επιτόπου είναι σημαντική ε, και ε, το Αφγανιστάν ε, υπήρξε μία βασική βάση ε, για τις επεμβάσεις μας ε, και μπορέσαμε να καταρτήσουμε την πυραμίδα προαγωγών της αστυνομίας στο Αφγανιστάν και ε, υπάρχει και ένα σκέλος το οποίο προωθεί το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών για να μπορέσουμε να προς ε, ε, ε, την τις εξελίξεις. Τώρα στην Αμερική το Υπουργείο Εξωτερικών, το State Department είναι υπεύθυνο για, τις, για την εκπαίδευση εις το Ιράκ, αλλά νομίζω ότι έχουν αντιληφθεί και αυτοί πλήρως ότι πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι, έχουμε μία πολύ στενή συζήτηση με το, τις Ηνωμένε Πολιτείες προσπαθώντας να αποφύγουμε τις επικαλύψεις και να καταλήξουμε από κοινού σε μια κοινή άποψη για το τι χρειάζεται για να αναπτυχθεί η αστυνομία στο Ιράκ και πώς θα μπορούμε να προχωρήσουμε από εκεί. Ένα άλλο μάθημα το οποίο αποκομίσαμε από αυτή την ε, αποστολή είναι η συνεργασία με τους άλλους Ευρωπαίους και την αντιπροσωπεία στο Ιράκ γιατί από όλες τις αποστολές αυτή ε, συνεργάζεται καλύτερα με το Ιράκ Ε, έχει έρθει ένα συνάδελφό σας, λέει ε, ο κύριος Γκάλερ, αλλά χωρίς μικρόφωνο. Ουσιαστικά οι αντιπροσωπείες αυτές είναι πολύ περιορισμένες. Πρόκειται για ένα άτομο μόνο, μάλιστα επί του προκειμένου ε, μία κυρία. Λειτουργούν πολύ καλά, προσπαθούμε να την βελτιώσουμε, αλλά αυτό είναι το βασικό θέμα ε, στο σημείο αυτό. Βέβαια, ενώ η κατάσταση ασφαλείας έχει βελτιωθεί, ε, είναι κακή και ουσιαστικά είναι χειρότερη από το Αφγανιστάν, πράγμα το οποίο εμποδίζει την ελευθερία κινήσεως και τη δυνατότητα να έχουμε αλληλεπίδραση ε, με το με τους συναδέλφους στο Ιράκ και να μπορέσουμε να επιτύχουμε και να προχωρήσουμε πολύ επί Όπως ξέρετε όμως ε, υπάρχουν εξελίξεις στο Ιράν που δεν ξέρουμε ποια θα είναι η έκβαση μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την αποστολή μας και τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την εντολή που έχει λάβει και μέχρι στιγμής πρέπει να πούμε ότι κάνουμε ό,τι μας είναι δυνατόν αλλά δεν υπάρχει μία γραμμική πρόοδος όπως θα έπρεπε αλλά όπως σας είπα είπα ε, κινούμεθα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον το οποίο βέβαια επηρεάζει και την ε, ε, απόδοση των κινήσεών μας και είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ιδιαιτέρως ένα βασικό στοιχείο το οποίο δεν υπάρχει είναι η συμφωνία με τους Ιρακινούς. Διότι στο Ιράκ αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι πρέπει να δώσουμε ε, στα μέλη της αποστολής ε, ασυλία από τις Ιρακινές αρχές, αλλά ότι με τις πινακίδες των αυτοκινήτων είναι εύκολο να μπει κανείς στην πράσινη ζώνη και αυτό είναι βέβαια το πιο ουσιαστικό σημείο ανασφαλείας ε, στο μηχανισμό. Πρέπει λοιπόν να συνεργαζόμαστε με την αντιπροσωπεία είτε για να βελτιώσουμε την απόδοσή της είτε για να προσθέσουμε κάτι το οποίο λείπει. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις τις οποίες ήθελα να κάνω πέραν αυτών που σας είπε ο Λάσλο ο και τώρα περιμένω με ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Όπως είπατε η αποστολή ξεκίνησε το 2005. Αυτό που υπάρχει τώρα είναι κάτι το νέο και γι' αυτό παρουσιάζει πολλές προκλήσεις. Και νομίζω ότι οι αρχές του Ιράκ χρειάζονται την αποστολή αυτή υπάρχουν ανάγκες για βελτιώσεις ιδιαίτερα στο θέμα της απονομής της δικαιοσύνης και σε σχέση κυρίως με τα ποινικά. Τρεις ερωτήσεις. Η συμφωνία η εταιρική και η συμφωνία συνεργασίας, τι ακριβώς συμβαίνει. Δεύτερο θέμα είναι η κατάσταση των, ε, ε, των φυλακών στο Ιράκ. Είναι μια γνωστή κατάσταση όχι καλή και διαρωτώ αν έχει υπάρξει ένα νέο νομικό πλαίσιο, αν σέβονται τα ελάχιστα επίπεδα τα οποία είναι αποδεκτά στην Ευρώπη και λοιπά. Και η τρίτη ερώτησή μου uh, I believe we, we put all the question Λοιπόν, σε σχέση τώρα με τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά ή τα επαγγελματικά τέλη, δεν ξέρουμε τι είπε η Πρόεδρος, περιμένω απαντήσεις. Η κυρία Κοπά, σας ευχαριστώ και τους δύο, λέει η κυρία Κοπά, για τις ε, παρουσιάσεις σας. Ακούγοντάς σας να μας εξηγείτε την αποστολή αυτή. κατανοεί κανείς τη δράση σας, όπως η ενίσχυση του κράτους δικαίου, η εκπαίδευση των αστυνομικών αρχών κτλ. Σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα στο Ιράκ, τι ακριβώς γίνεται. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά την ορατότητα της συγκεκριμένης αυτής αποστολής στο Ιράκ και την αποδοχή της από τον λαό του Ιράκ. Τώρα μετά την απόσυρση των ξένων στρατευμάτων γνωρίζετε ότι υπάρχει η πολιτική βούληση και υπάρχει η ικανότητα των Ιρακινών αρχών να αναλάβουν ε, δράση, να καλύψουν τα κενά. Και τέλος ε, με μια πιο τεχνική ερώτηση. Σύμφωνα με την εντολή της αποστολής, εκπαίδευση, κατάρτιση, την οποία παρέχουν λέγεται τα κράτη-μέλη λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα διάφορα κράτη-μέλη. Πόσο έχετε επηρεαστεί στα πλαίσια της συμμετοχής στην αποστολή σας και της αποτελεσματικότητάς της. Ο κ. Γκάλα. Ευχαριστώ. Περιμένω όμως να βάλετε τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Καταρχήν ε, χαίρομαι ε, διότι πριν ακόμη θέσω τις ερωτήσεις ορισμένες είχαν ήδη απαντηθεί ότι για το πόσο προχωρούν ε, οι σχέσεις με την Αμερικανική Αποστολή και χαίρομαι που είναι τόσο καλές και ότι συνεχίζεται αυτό το οποίο είχε θεσπιστεί προηγουμένως. Αυτό με χαροποιεί ιδιαιτέρως. Επανέρχομαι όμως διότι το αναφέρατε και πριν στο θέμα του πώς ε, είναι η συνεργασία, πώς δηλαδή διαμορφώνεται η συνεργασία με τους Αμερικανούς. Μπορείτε να τους πείσετε ή λένε εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας, αυτό θα εφαρμόσουμε και αν κάτι περισσέψει κάντε ό,τι μπορείτε. Πώς δηλαδή ε, γίνεται αυτός ο συντονισμός, διότι μπορώ να αντιληφθώ ότι επιτόπου τόπου ενδεχομένως δεν υπάρχει ο σωστός μοχλός. Πρέπει να υπάρξει μία πολιτική συνεννόηση και απόφαση είτε στις Βρυξέλλες με την Αμερικανική ε, Περεσβεία είτε με, ε, στην Ουάσιγκτον. Τι γίνεται στο θέμα της, ε, της αστυνομίας. Οι βλέψεις των Αμερικανών και οι απόψεις τους συνάδουν με με τις δικές σας ή ο καθένας έρχεται από το δικό του κόσμο και δεν υπάρχει μία συμφωνία μεταξύ των δύο. Ένα άλλο θέμα είναι ότι μου είπατε ότι ήδη λειτουργούμε από το 2005 αλλά στην αρχή ε, ε, εκ Βρυξελών και αντιλαμβάνομαι ότι διάφορα κράτη προσέφεραν ορισμένες δυνατότητες και καταρτίστηκαν ε, οι διάφοροι μηχανισμοί. Πώς λοιπόν σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της εκπαιδεύσεως ε, πόσο μπορούμε να τα αξιολογήσουμε επί τόπους. Δηλαδή, ο Τάδε, ο οποίος ήταν εδώ το 2005 και το 2006 και τώρα κατέχει αυτή τη θέση, έχουμε την εντύπωση ότι τα έχει καταφέρει και κατάλαβε περί σε πρόκειται. Πώς αξιολογείται λοιπόν τις επιτυχίες μίας εκπαιδεύσεως η οποία έχει γίνει εκτός της χώρας. Θέλω επίσης να ρωτήσω, δραστηριοποιήστε και στην Κουρδία δική πλευρά ή μόνο ή στον κεντρικό χώρο. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ, ο κύριος Τέχο. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για τις πάρα πολύ καλές παρουσιάσεις. Σας θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η εμπειρία σας από τη βάση, δηλαδή οι απλή πολίτες, ο άμαχος πληθυσμός σας εμπιστεύεται, πώς σας αντιμετωπίζει και ιδίω τι γίνεται ε, στις σχέσεις με τις ε, αρχές της χώρας, πώς αντιμετωπίζουν. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εθνικές συγκρούσεις. Βλέπετε και, μεταξύ, και στους κόλπους της αστυνομίας ε, να υπάρχει ε, κάποια αντιπαράθεση ενδεχομένω. Τέλο πάντων οι διάφορες ε, εθνότητες αντιπροσωπεύονται ισομέρό στα σώματα ασφαλείας. Τι γίνεται λοιπόν στο δικαστικό σώμα αλλά και στην αστυνομία. Którą Καταρχάς θέλω να πω ότι εκτιμώ ε, πάρα πολύ τη δουλειά που κάνετε επί στο Ιράκ. Πρέπει να σας πω ότι στη δική μου σταδιοδρομία για τρία χρόνια ήμουν ε, αρμόδιος ε, για την πολωνική μεραρχία εκεί, είχαμε πάει και στη, σε διάφορες περιοχές. Γνωρίζω την κατάσταση επιτόπου πολύ καλά και ξέρω πόσο δύσκολη και επικίνδυνη είναι η αποστολή εκεί. Γι' αυτό και πραγματικά τρέφω περιόριστο σεβασμό στον καθένα και στην καθεμία που βρίσκεται επιτόπου στο Ιράκ, γιατί γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν. Έρχομαι σε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Τρία τον αριθμό. Πρώτο ερώτημα. Είναι γενικό και το απευθύνω προς τον ε, κύριο Πρέσβη. Ποια είναι η αξιολόγηση ε, που μπορείτε εσείς να κάνετε της κατάστασης στο Ιράκ. Είπατε ότι βλέπετε εδώ και κάποιες ημέρες ε, κάποια αλλαγή, ότι αυτό κάπως αυτή την εντύπωση έχετε αποκόμιση ότι κάπως αλλάζουν τα πράγματα. Πώς μια κατεύθυνση όμως, αυτό θα ήθελα να μας πείτε με λίγο μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Τα επόμενα δύο ερωτήματά μου ε, απευθύνονται στον στρατηγό Χούσαρ. Το πρώτο, έχει εγκρίνει το νέο ε, ποινικό και αστικό κώδικα το Ιράκ. Γιατί ξέρω ότι είναι μια πηγή, ε, είναι ένα διαφιλονικούμενο ζήτημα εκεί. Δεύτερο ερώτημα το προσωπικό που έχετε στη διάθεσή σας. Νομίζω είπατε 37 άτομα. Στην Βαγδάτη και στην Μπάσρα είπατε 6 άτομα, αν θυμάμαι καλά. Δεν νομίζω ότι αντικατοπτρίζουν οι αυτή αυτοί τη δυνατότητα που θα μπορούσε ε, να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είναι πολύ, πιο πολύ άριθμο το προσωπικό εκεί. Το θέμα είναι ότι μετά την απόσταση των στρατευμάτων πρέπει να βοηθήσουμε τους Ιρακινούς και σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση λοιπά. Αυτά τώρα ήταν ε, μόνο εξαγγελίες, ε, δηλώσεις ή πραγματικά έχουμε παρουσία επιτόπου. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί που λέτε ότι είναι επιτόπου, τι είδους εμπειρογνώμονες είναι, πού ειδικεύονται στην εκπαίδευση των ε, αστυνομικών, των ανώτερων όμως αξιωματικών αστυνομίας. Τι ακριβώς κάνουν εκεί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για εμάς. Και θα ήθελα να μου πείτε, γιατί νομίζω ότι κάποιες χώρες έχουν πάρει πιο σοβαρά την αποστολή αυτή από τις άλλες. Κυρία Κρόμπερ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να έρθω στις εθνωτικέ συγκρούσει, αλλά πιο πολύ ε, στις θρησκευτικέ σχεσεις δηλαδή μεταξύ των Σιητών. Επηρεάζει αυτό τις δικές σας ε, δυνατότητες να φέρετε σε πέρας με επιτυχία την αποστολή σας. Βλέπετε μήπως τίποτα ανησυχητικά δείγματα για κάποιον εμφύλιο πόλεμο ενδεχομένω. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ιράν και την Ιρανική επιρροή στο Ιράκ. Αυτό επηρεάζει ε, κάπως τον, ε, το δικό σας έργο. Μπορείτε να μας πείτε τι είδους επιρροή έχει αυτή τη στιγμή το Ιράν στο Ιράκ. Στάνσκι. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Χαμπέρ. Έχουν τεθεί πολλές ερωτήσεις, περιμένω τα σχόλιά σας. Μια απλή ερώτηση. Θα ήθελα να μάθω ποιος είναι ο ρόλος ε, των τέος μελών του κόμματος Μπαθ. Παίζουν κάποιο ρόλο, περιορίζεται ο ρόλος τους. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς. Υπάρχει εμπλοκή τους στην πολιτική ζωή, έχετε επαφές μαζί τους. Λοιπόν, ποιος θέλει να απαντήσει πρώτος, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Χούτσαρ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η εταιρική σχέση είναι μια καλή ευκαιρία. Ελπίζω ότι αποδεικνύει και την πολιτική βούληση της Ιρακινής πλευράς. Δεν είναι αυστηρά σε πολιτικό επίπεδο. Η συμμετοχή μας είναι τεχνική Ελπίζουμε όμως ότι με τη νέα αυτή συμφωνία θα αυξηθούν οι δυνατότητες τις οποίες έχουμε και θα βελτιωθεί και το επίπεδο, σε, και το επίπεδο αν θέλετε, αξιοπιστίας της αποστολής μας και σε επίπεδο πρωτοκόλλου η αποστολή μας θα προβιβαστεί κατά κάποιο τρόπο σχετικά με τις φυλακές μετά από εμπειρίες που είχαμε επιτόπου, τα επίπεδα στις φυλακές ποικίλουν. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν, θα έλεγα, κάποια επίπεδα επαγγελματισμού. Από την άλλη, τα στοιχεία και τα ίχνη του προηγούμενου αυταρχικού καθεστώτος και κάποιες άλλες τοπικές παραδόσεις δημιουργούν προβλήματα και σήμερα. Εμείς τους εκπαιδεύουμε, τους δεσμοφύλακες ε, στα ευρωπαϊκά επίπεδα, διδάσκουμε ε, συστήματα διαχείρισης και βελτίωσης ε, της λειτουργίας των φυλακών, συστήματα ελέγχου της λειτουργίας των φυλακών, διαχείρισης γενικότερα των σοφρονιστικών θεσμών. Για τη δικαστική εξουσία είμαστε σε συνεχή επαφή με το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και την Ανώτατη Εισαγγελία είναι αρκετά καλά εκπαιδευμένοι. Έχουν μεγάλη παράδοση δικαστική και νομοθετική. Στο Ιράκ πολλές δεκαετίες, αλλά χρειάζονται καλύτερη οργάνωση, καλύτερη θα έλεγα διαχείριση έχουν να ασχοληθούν όμως και με νέου είδους εγκληματικές δραστηριότητες ε, όπως καταχρήσεις κτλ ε, τις οποίες δεν γνώριζαν στο παρελθόν. Σχετικά τώρα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουμε δύο συναδέλφους που ασχολούνται με το θέμα αυτό και στόχος τους είναι να δίδουν συμβουλές στους εκπαιδευτές έτσι ώστε ε, να υπογραμμίζουν οι εκπαιδευτές τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ε, διάστασης των φύλων. Εμείς ε, οργανώνουμε μαθήματα, διδάσκουμε τους, αυτούς οι οποίοι καλούνται να διδάξουν με τη σειρά τους Πάντως υπάρχουν και άλλες οργανώσεις ε, οι οποίες ασχολούνται στη χώρα με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως το UNDP. Τώρα, για την εικόνα που έχουμε και την πολιτική βούληση να συνεχίσουμε. Οι Ιρακινοί ομολογοί μας θέλουν να συνεχίσει η αποστολή η εκπαίδευση την οποία παρέχουμε και θέλουν να ενσωματώσουν την τεχνογνωσία την οποία τους μεταφέρουμε. Έχουμε μια καλή προοπτική σχέση μαζί τους και οι εμπειρίες που μεταφέρουμε είναι χρήσιμες. Υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες ε, συνεισφέρουν στην αποστολή μας. Δεν θα τις απαριθμίσω. Πάντως άνω των 10 χωρών συμμετέχουν. Κάποιοι από αυτούς είναι σύμβουλοι, κάποιοι από αυτούς έχουν έρθει με συμβάσεις δηλαδή, κάποιοι είναι αποσπασμένοι Έχουμε διαφορετικού τύπου επαγγελματίες, δικηγόρους, νομικούς μάλλον, αστυνομικούς. Έχουμε και κάποιους υπεύθυνους σοφρονιστικών συστημάτων. Regarding the US, uh, uh, the US uh, uh, cooperation with the United States, uh, um, it, it works in a way that we meet regularly. Um, uh, uh, uh, and discuss our plans. Εμείς προσπαθούμε να προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας στις δυνατότητες ανάλογα και με τις τοπικές ανάγκες. Συνεργαζόμαστε και με άλλες χώρες. Χθες είχαμε, θα έλεγα, οργανώσαμε μάλλον χθες συγκεκριμένα σε συνεργασία με τους Αμερικανούς ένα σεμινάριο για τις εκλογικές διαδικασίες. Και η ανταλλαγή εμπειριών με τους Αμερικανούς ήταν πολύ χρήσιμη. Ε, for criminal investigation, tactical investigation, and we asked our American colleagues. Um, και σε επίπεδο ανακριτικών δυνατοτήτων έχουμε συνεργαστεί με τους Αμερικανούς και τους έχουμε ζητήσει να πάρουν μέρος στις διαδικασίες εκπαίδευσης. Η συνεργασία μαζί τους είναι καλή και σε τεχνικό επίπεδο. Οι διαπραγματεύσεις δεν ασχολούνται με το αν θα υπάρξει δυνατότητα για κάποιες οργανώσεις να κάνουν κάποιες ε, δράσεις εκπαιδευτικές. Υπάρχει μια κατανομή αρμοδιοτήτων, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν στο Ιράκ και γι' αυτό νομίζω υπάρχει χώρος και για τους Αμερικανούς και για μας και μαζί μπορούμε να πετύχουμε. Οι Αμερικανοί ας πούμε ασχολούνται με θέματα με τα οποία εμείς δεν ασχολούμεθα, όπως εκπαίδευση σκύλων αστυνομικών. The content of these, uh, these uh, specialized uh, police training, uh, but it wouldn't, uh, wouldn't uh, uh, uh, collude or clash with... Προσπαθούμε πάντως ε, να, μην, ε, να συντονιζόμαστε και να μην υπάρχουν επικαλύψεις ανάμεσά μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άσχετο αν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν θέματα επαγγελματικής κατάρτισης είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο δικό μας. Σχετικά με το λεγόμενο benchmarking των διαδικασιών κατάρτισης. Έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα πλήρες ελέγχου των πεπραγμένων. Εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τις γνώσεις τις οποίες παίρνουν από τις συναντήσεις μαζί μας και πώς τις εφαρμόζουν επαγγελματικά. Φυσικά όλα αυτά δεν είναι πάρα πολύ εύκολα Είναι δύσκολο, όπως είπα, επειδή είναι μεγάλη χώρα να ταξιδεύει κανείς ή να φέρνει σε μία συγκεκριμένη περιοχή κόσμο από άλλες. Αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε να οργανωθούμε, ε, κάνουμε προσκλήσεις σε συναντήσεις εκ των υστέρων μετά το τέλος μιας κάποιας διαδικασίας κατάρτισης, έτσι ώστε να συλλέξουμε τις εμπειρίες από τη χρήση της. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα παραδοσιακά μέτρα που χρησιμοποιούνται σε, άλλες, σε άλλους τομείς, αλλά έχουμε ένα σύστημα το οποίο παρακολουθεί, εν πάση περιπτώσει, το τι ακολουθεί των διαδικασιών κατάρτισης. Για το κουρδικό, για την κουρδική περίπτωση μάλλον, έχουμε ένα γραφείο στο Αρμπίλ, Στο Κουρδιστάν η κατάσταση ασφαλείας είναι πολύ καλύτερη και μπορούμε να μετακινούμεθα με μεγαλύτερη ευκολία. και εκεί ε, κάνουμε σεμινάρια για τα δικαστήρια, τα περιφερειακά της κουρδικής περιοχής. Η κατάσταση ασφαλείας μετά την απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων Είναι πολύ δύσκολο να κρίνει κανείς τόσο γρήγορα, ένα μήνα μετά δηλαδή περίπου από την αποχώρηση των Αμερικανών. Εγώ το βλέπω σε επίπεδο πρακτικό και όχι πολιτικό βέβαια. Νομίζω ότι η κατάσταση ασφαλείας στη χώρα τουλάχιστον σε επίπεδο λειτουργικό θα έλεγα, επιχειρήσεων μάλλον, δεν έχει χειροτερεύσει. Το σύστημα γενικά ελέγχου των συνθήκων ασφαλείας και τα λοιπά δεν έχει καταρρεύσει. Προφανώς και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα Υπάρχουν επίσης ε, κοινοτικά προβλήματα, ε, κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα ανάμεσα στις κοινότητες, εθνοτικά προβλήματα, αλλά δεν παρεμποδίζουν, θα έλεγα, τις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες. στις εκπαιδευτικές μας δράσεις. Υπάρχουν εκπρόσωποι δικαστές ε, και Σούνη και Σία. Λειτουργούμε σε ένα προστατευόμενο θα έλεγα περιβάλλον και ε, οι συγκρούσεις ε, όχι ότι δεν υπάρχουν αλλά τουλάχιστον δεν εκδηλώνονται. σχετικά με την ποινική νομοθεσία είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και επηρεάζει και το ποινικό κομμάτι και το αστικό κομμάτι, νομοθετικά εννοώ. Δεν έχουν αλλάξει ακόμα πάρα πολλά πράγματα. Ισχύουν οι παλαιές νομοθετικές ρυθμίσεις, από τη δεκαετία του 50 ισχύουν ή από την εποχή του καθεστώτος Σαντάμ. Έχουν γίνει πρακτικές προτάσεις για αλλαγές, αλλά τα βασικά ισχύοντα κείμενα, οι βασικοί ισχύοντες νόμοι είναι οι ίδιοι. Υπάρχει και μια επιτροπή ελέγχου του κράτους δικαίου στη Βαγδάτη. Συμμετέχουμε και εμείς με Ιρακινούς φυσικά συναδέλφους κυρίως. Ε, την τελευταία συνάντηση ενημερωθήκαμε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Μεταρρύθμισης της Νομοθεσίας τις ε, προτάσεις που έχουν γίνει και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες αλλαγής του ποινικού κώδικα, σαν παράδειγμα. Υπάρχουν πράγματα λοιπόν που γίνονται, υπάρχουν πράγματα που εξελίσσονται και στον τομέα το νομοθετικό, Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, είναι περίπλοκη αυτή που ακολουθείτε, αλλά είναι κάτι που προχωρά. Όπως είπα, οι φιλετικές διακρίσεις της Ιρακινής κοινωνίας δεν είναι κάτι το οποίο καλούμε εγώ να σχολιάσω. Όπως και άλλα πολιτικά περισσότερα θέματα, όπως οι σχέσεις του Ιράκ με το Ιράν. Εμείς δεν το βλέπουμε αυτό στην καθημερινή μας πρακτική, αλλά σας είπα ποια είναι η προοπτική μας, είναι περιορισμένη, συγκεκριμένη. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να έδωσα κάποιες απαντήσεις. Οι ερωτήσεις σας ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Τίποτα άλλο. Ο κύριος Χαμπέρ. Νομίζω ότι οι περισσότερες ε, ερωτήσεις σας ε, ουσιαστικά απαντήθηκαν από τον Λάσλο και εγώ δεν έχω να προσθέσω πολλά από την οπτική γωνία των Βρυξελών και μην έχοντας την εμπειρία επιτόπου στο Ιράκ, αλλά θα κάνω μερικές παρατηρήσεις οι οποίες ίσως σας ενδιαφέρουν. Σε αυτή την αποστολή, όπως και σε όλες τις άλλες, εκτός δύο, ουσιαστικά ε, έχουμε εμπλακεί σε έναν τομέα ασφαλείας σε έναν τομέα, δηλαδή στην ε, ε, μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας. Ε, και αυτό έχει αναλυφθεί κατά μεγάλο μέρος από τους Αμερικανούς και οι Αμερικανοί να γνωρίζουν ότι έχουμε καλύτερη παιδεία στην εκπαίδευση της αστυνομίας, τουλάχιστον στην κορυφή της πυραμίδας για εθνική αστυνομία από ό,τι στην Αμερική και αυτό απεδείχθη ήδη από την κατανομή ε, των εργασιών που είχε γίνει στην προηγούμενη αποστολή στο Αφγανιστάν. Οπότε ε, όλα αυτά ίσως ε, έχουν κατακριθεί σε πολλά επίπεδα, αλλά τα δύο επίπεδα τα οποία εμείς ε, αντιμετωπίζουμε είναι άπαξ και εκπαιδεύσουμε τους αστυνομικούς πώς θα πληρωθούν, το οποίο ήταν πρόβλημα στο Αφγανιστάν, όχι όμως ελπίζουμε στο Ιράκ που είναι μία πλούσια χώρα και πώς θα διεκπεραιώνει αυξάνεται η δικαιοσύνη, διότι αν η αστυνομία κάποια στιγμή δεν παραπέμπει τα θέματα στην δικαιοσύνη, τότε είναι μία κρυφίως ε, τοποθετημένη ε, στρατιωτική δύναμη. Προσπαθούμε λοιπόν πάντοτε να ε, τονίσουμε περισσότερο το θέμα της ε, ε, αστυνομίας και των φυλακών εφόσον ο Λάσλο προέρχεται από το σοφρονιστικό σύστημα της Ουγγαρίας και να αναπτύξουμε τη συνεργασία μεταξύ αστυνομίας και δικαιοσύνης. Δηλαδή να υπάρχει ε, η δυνατότητα και να το γνωρίζουν όλοι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μεταβιβαστεί από τον έναν στον άλλον αρμοδιότης και υπάρχουν και περιορισμοί ε, οι οποίοι εσείς μπορείτε να επιφέρετε ε, σε αυτήν την δομή πώς ε, πρόκειται να προωθηθεί και η περισσότεροι ε, είναι ε, είναι ε, όντως έμπειροι από τους εκπαιδευτές αλλά ε, ένα άλλο θέμα είναι ότι όταν κινείστε με τεθεροκισμένα οχήματα από την πράσινη ζώνη προς τα έξω αυτό είναι μια εικόνα για τους πολίτες την οποία βλέπουν εδώ και 8 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή μια εμφανής ευρωπαϊκή παρουσία. Αυτή υπάρχει μόνο μέσω του, είπα, του υπευθύνου ε, και ελπίζουμε ότι θα αναπτυχθεί. Ε, επειδή όμως στο Ιράκ υπάρχουν τα οχήματά μας, επειδή μπορούν οι δικοί μας να μιλήσουν με τους πολίτες ε, και στα θέματα όπου μπορούμε να επέμβουμε ε, σε άλλες χώρες μας βλέπουν αλλά στο Ιράκ αυτό δεν συμβαίνει και πιστεύω ότι για τα περαιτέρω η πληροφόρησή μου είναι όπως ε, και η δικιά σας από εφημερίδες, από την Γιάννα και αυτά είναι μέρος της κατανομής εργασίας την οποία έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι η ερώτηση αυτή θα έπρεπε να τεθεί στην Γιάννα. Όλοι βέβαια γνωρίζουμε ότι υπάρχει ε, ένας ε, κίνδυνος να υπάρξει και πάλι μία αναζωπήρωση των διαμαχών μεταξύ ε, των διαφόρων πλευρών και το ενδιαφέρον που αισθάνονται οι Ιρακινοί βασίζεται στο να μπορέσει να γίνει το δικό τους και γι' αυτό απεσύρθη η αποστολή του ΝΑΤΟ. Εμείς αυτή τη στιγμή ε, δεν έχουμε μία αποκρισταλωμένη θέση, αλλά ε, έχουμε μία ταυτότητα πολύ πιο σαφή από ότι οι Αμερικανοί και έτσι έχει εξελιχθεί η κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία βιώσιμη ρύθμιση για τις δυνάμεις που έχουμε αναπτύξει επί τόπου. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Αν όχι, Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και τους δύο για την ενδιαφέρουσα και πολύ ειλικρινή ε, παρουσίαση. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολη η δουλειά σας, κάνετε ε, πολλές προσπάθειες ε, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την ισότητα των φύλων και για να ε, μπορέσει να υπερισχύσει η ποινική δικαιοσύνη που είναι κάτι που χρειάζεται σε όλες τις χώρες αλλά αισθάνομαι ότι τουλάχιστον στο Ιράκ έχει γίνει γίνει καλή δουλειά ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. colleagues allow me to invite αγαπητοί συνάδελφοι, να προσκαλέσω τον επόμενό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Θεότορ Βίνκλερ, πρέσβη. Παρακαλώ. Okay, we can continue the... Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο της μερικής διάταξης. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρέσβη Βίνκλερ. Διευθυντή του Κέντρου Δημοκρατικού Ελέγχου των Ανώπλων Δυνάμεων της Γενέφης. Δίκαφ θα το λέμε εν συντομία του κέντρου, από εδώ και πέρα. Το DICAF ξέρετε ότι είναι ένα διεθνέ ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 2000 κατόπιν πρωτοβουλίας της Ελβετίας με στόχο να στηρίζει την ε, λογοδοσία στον τομέα της ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλω να σας υπενθυμίσω πόσο χαιρόμαστε που το DICAF εκ μέρους ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει διενεργήσει σημαντικές μελέτες ε, για το θέμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου της κοινή ε, πολιτικής ασφάλειας και άμεσα του κοινοβουλευτικού ελέγχου, της ασφάλειας, τα συστήματα πληροφοριών, intelligence και αυτά ήταν απλά κάποια παραδείγματα. Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Δίνω το λόγο στον πρέσβη. Euh, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω πολύ σύντομα το Κέντρο Δημοκρατικού Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων, το ΔΙΚΑΦ. Και θα σας ε, εκθέσω τις δραστηριότητές μας ή μέρος αυτών. Όπως ε, προείπε η πρόεδρός σας, το ΝΤΙΚΑΦ αποτέλεσε πρωτοβουλία της ελβετικής κυβέρνησης τον Οκτώβριο του 2000, ένα διεθνέ ίδρυμα. Από νομικής πλευράς λοιπόν είναι μη κυβερνητικό, μη κρατικός οργανισμός, ωστόσο τα μέλη μας είναι κράτη. Είμαστε δηλαδή κυβερνητικός, διακυβερνητικός, μη κυβερνητικός οργανισμός ή κάτι από όλα αυτά κάτι μεταξύ διεθνούς οργανισμού και μη κυβερνητικής οργάνωσης. Σήμερα ε, αριθμούμε 64 μέλη από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 130 περίπου είναι οι συνεργάτες μας από ολόκληρο τον κόσμο. Ο προπολογισμό μας είναι 30 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, 25 εκατομμύρια ευρώ. Αντιστοίχω και η ελβετική ε, κυβέρνηση συνεισφέρει με το 45% και το υπόλοιπο 55% το καλύπτουν τα άλλα κράτη-μέλη, αλλά οι εισφορέ είναι εθελοντικέ. Η συμμετοχή είναι εθελοντική. Η αποστολή μα δεν είναι μόνο δημοκρατικό έλεγχο ε, των ένοπλων δυνάμεων, αλλά ευρύτερα η καλή διακυβέρνηση και η μεταρρύθμιση τομέα τη ασφάλεια. Αν με επιτρέπετε τώρα να περάσω στα αγγλικά. Forces, but also with the police, with border guards, intelligence agencies. Με τις παρτιωτικές δυνάμεις, ιδιωτικές ε, δυνάμεις και εταιρείε ασφαλείας και με άλλες μορφές κρατικές αρχές ή άλλες ε, προσπαθούμε να συνεργαστούμε. Θα σας αναφέρω κάτι πολύ σοβαρό και σημαντικό και σε αυτά τα πλαίσια. Μηχανισμοί ελέγχου. Υπουργικοί, υπουργικές δομές, αλλά κυρίως ε, κοινοβουλευτικός έλεγχος, που είναι πάρα πολύ σημαντικός, αλλά και συνεργασία με την κοινότητα των πολιτών και με το δικαστικό σώμα. Τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Πρώτα απ' όλα, σε πολλές χώρες που μετάβαση ο τομέας ασφάλειας είναι σαν κράτος εν κράτη. Δηλαδή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως δημοκρατία όπου υπάρχει κράτος δικαίου. Κάποιες φορές δεν υπάρχει καν ασφάλεια. Παρομοίως, έχουμε αυτή την, το κρατικό μονοπόλιο των ενόπλων δυνάμεων που έχει ε, καταρρεύσει. Άρα δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ειρήνη όπως βλέπουμε με το Ισραηλινο-Παλαιστινιακό πρόβλημα. Πόσο δύσκολο είναι να ελεγχθεί η βία, παρότι είναι ένα θέμα πρωταρχικής σημασίας. Τρίτο παράδειγμα. Μετά τις συγκρούσεις, ε, πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένας ε, λειτουργικός τομέας ε, ασφάλειας που θα είναι διαφανώς οργανωμένος, δημοκρατικά νομιμοποιημένος και ελεγχόμενος αυτό είναι προϋπόθεση για ειρήνη, ασφάλεια και κράτος δικαίου. Δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη χωρίς την προϋπόθεση αυτή. Εάν δούμε ευρύτερα τα πράγματα, θα δούμε ότι η πείνα και η φτώχεια συνδέονται πολύ στενά και με τη δημιουργία δημοκρατικώς νομιμοποιημένων ε, δομών ασφάλειας. Χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Κανείς δεν μπορεί να επενδύσει σε μια μπόλεμη περιοχή ή δεν θέλει να το πράξει. Η ασφάλεια βέβαια δεν θα πει μόνο αστυνομική παρουσία στους δρόμους, αλλά σημαίνει πώς μπορούμε συγκεκριμένα να οργανώσουμε την κοινωνία με διαφανή τρόπο με δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία. Η πείνα είναι ένα πρόβλημα. Όταν κάποιο το στομάχι είναι άδειο, τίνει πιο εύκολα να πιάσει ένα καλάσνικο στο χέρι. Άρα η ασφάλεια έχει να κάνει και με τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Πρέπει να δούμε λοιπόν διάφορε πτυχέ για την ε, διαχείριση και την πρόληψη των συγκρούσεων και την ανοικοδόμηση μετά από ε, σύγκρουση πολλές προκλήσεις και πρέπει να αναπτύξουμε σχετική πολιτική. Είναι ένα τρίγωνο λοιπόν, κράτος δικαίου, ανάπτυξη, ασφάλεια. Και πάνω σε αυτό το τρίγωνο, μέσα σε αυτό το τρίγωνο λειτουργούμε και εμείς, το DICAF, με τριπλή αποστολή, πάνω σε τρία επίπεδα. Πρώτο επίπεδο, στηρίζουμε τη διεθνή κοινότητα στις προσπάθειες ανάπτυξης μιας συνεκτικής στρατηγικής. Για το SSG και το SSR. Το ΔΙΚΑΦ είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος του ΟΗΕ. Συνεργάζεται και με το ΙΝΟΑΣΕ και με άλλους σημαντικούς ε, οργανισμούς ε, όπως και η Αφρικανική Ένωση, η ΑΣΕΑΝ και άλλοι οργανισμοί. Αλλά, αυτό που με φέρνει και στις Βρυξέλλες βέβαια, Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργασία. Δεύτερο επίπεδο, ανάλυση το κέντρο συλλέγει, αναλύει, ε, διασμοσιεύει καλές πρακτικές ε, και διδάγματα που έχουμε αντλήσει σε αυτούς τους τομείς. Χιλιάδες μελέτες και εγχειρίδια δημοσιεύουμε κάθε χρόνο, τα οποία έχουν μεταφραστεί, μεταφράζονται σε πάνω από 45 γλώσσες. Άρα δεν καλύπτουμε μόνο ε, τις χώρες ε, της επίσημης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής κάνουμε μεταφράσεις και σε άλλες γλώσσες. Το DICAF ε, είναι προσανατολισμό στις επιχειρήσεις. 400 ε, projects επιτόπου ε, διευθύνουμε με πολύ μεγάλη έμφαση στη δημιουργία δυνατοτήτων υποδομών και την τοπική ιδιοκτησία, το local ownership. Θα σας δώσω κάποια παράδειγμα, δείγματα του επιχειρησιακού μας έργου. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βοηθήσουμε την, την νησιακή κυβέρνηση να ξεπεράσει τα κληροδοτήματα της κυβέρνησης Μπεναλή και της δικτατορίας. Ένα μέλος του ΝΤΙΚΑΦ από το καλοκαίρι βρίσκεται και αναπαράσχει βοήθεια στη διάδοχη κυβέρνηση. Και χθε συγκεκριμένα, ε, μάλλον ένα χρόνο από χθε, ξεκίνησαν αυτές τις προσπάθειες και τώρα έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Έχουμε διάφορα μνημόνια συνεργασίας και συνεννόησης με πολλά υπουργεία, ιδίω του εσωτερικών και της δικαιοσύνη, αλλά και του προεξωτερικών και άμυνα στην Τινησία. Προσπαθούμε λοιπόν να βοηθήσουμε στη μεταρρύθμιση πολλών πτυχών στην τινησιακή πραγματικότητα, από το θέμα των δύο φύλων, πρακτικά ζητήματα, κράτηση, σύστημα κράτηση ε, κτλ. Ε, διαχείριση αρχείων ε, που έχει αφήσει πίσω τη κυβέρνηση Μπέναλη μηχανοργάνωση, κανονισμοί για την ε, δημόσια διοίκηση λοιπά. Θέλουμε να τα μεταφράσουμε δε και να υπάρχουν σε αραβικά, αγγλικά και γαλλικά όλα αυτά τα κείμενα και οι κώδικες. Επίσης προσπαθούμε να βοηθήσουμε την τρίτη πλέον σε ένα χρόνο κυβέρνηση να βρει το δρόμο της να δει τι μπορεί να κάνει, πώς να αντιμετωπίσει τα πολυσχεδή προβλήματα της χώρας. Και αυτό το πράττουμε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους εκπροσώπους της Επιτόπου, αλλά όχι μόνο και με τους εμπειρογνώμες εδώ επίσης, στο Μαρόκο, την Αίγυπτο, δραστηριοποιηθούμε, θα ελπίζουμε σύντομα και στη Λιβύη. Την επόμενη εβδομάδα είναι η πρώτη μας αποστολή εκεί. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις επίσης και στη Συρία και έχουμε γραφεία στη Ραμάλα και στη Βηρητό. Με πρωτοβουλία του ΑΣΕ δημιουργεί σαν με το λεγόμενο ISAD, που είναι μια μονάδα του Ντίκαφ και ενεργεί εξ ονόματος ε, της διεθνούς κοινότητας κάνει διάφορες αποστολές ε, παρακολούθησης επιτόπου, ιδίω ε, στην Αφρική αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ISAP προσπαθεί να αξιολογεί την κατάσταση σε διάφορες χώρες και έτσι να διευκολύνει τα προγράμματα συνεργασίας SSG-SSR. και να συμβάλλει στο συντονισμό των προσπαθειών. Και το ISAT και το DICAF Επίση ε, πολύ συχνά κάνουν αποστολέ εξ ονόματο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τονίσω και μια άλλη πλευρά. Υπάρχει μια υποεπιτροπή στην ISAT, ε, υποεπιτροπή που έχει και δικό της διοικητικό συμβούλιο, 14 ε, χώρες που είναι από τι βασικέ δωρητρίε χώρε και εκπροσωπούν βέβαια ο ΙΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, UNDPO κτλ. Αφρικανική Ένωση, Αφρικανική ε, Τράπεζα Ανάπτυξης ε, λοιπά. Είναι ένα σκόμβος διεθνούς συντονισμού. Και μπορεί να διεξαγάγει ταυτόχρονα πέντε αποστολές και στα γαλλικά και στα αγγλικά. Τρίτο παράδειγμα, στα Δυτικά Βαλκάνια. Το αντίκαυσε περιφερειακό επίπεδο είναι ο μεγαλύτερος πάροχος εμπειρογνωμοσύνης στο τομέα της αστυνομίας και της ε, και του συνοριακού ελέγχου. Έχουμε και στη Λιμπλιάνα ένα γραφείο και στο γραφείο στι Βρυξέλλε, βέβαια, γίνονται πολλά πράγματα, αλλά και από τη Λιμπλιάνα γίνονται επίση ε, πολλέ προσπάθειε. Ε, Σπαθούμε να εφαρμόσουμε τη σύμβαση τη Γενέβη. Εννέα χώρε ε, συνεργάζονται. Την Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυστρία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Η σύμβαση αυτή αποσκοπεί στο να υπάρξει επίπεδο συνεργασίας και συντονισμού ε, στην αστυνομία και στη συνοριοφυλακή, πέραν των συνόρων. Αυτή η σύμβαση λοιπόν PCC δεν είναι το μόνο που κάνουμε. Έχουμε και ένα πρόγραμμα ε, για την εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων στα Δυτικά Βαλκάνια. 40 συνεδριάσεις εμπειρογνωμών, υπουργικές συναντήσεις, σεμινάρια, εργαστήρια και άλλε συναθρήσει εμπειρογνωμόνων το χρόνο. Τώρα, εμείς από πλευρά Ελβετίας είμαστε μέλος του οργανισμού υλοποίηση για το Ταμείο Διεύρυνση για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από την πλευρά τη ε, Ελβετία. Έχουμε μια εξωτερική ανάθεση της, ε, των ε, πολυμερών προγραμμάτων αστυνομική συνεργασία που η Ελβετία το έχει αυτή την αρμοδιότητα την έχει μεταφέρει σε εμά, στον ΤΙΚΑΦ. Επίσης, για τη γραμματεία του κώδικα διοντολογίας ε, παρέχουμε τη σχετική υποστήριξη. Αυτός ο κώδικας έχει υπογραφεί από περισσότερες από 300 εταιρείε μέχρι σήμερα πάνω από το 95% αυτών που, ε, διεθνούν, που δραστηριοποιούνται διεθνώς. Δύο εκατομμύρια εργαζόμενοι. Προπολογισμό συνδυασμένο πάνω από 100 δις δολάρια. Και τα μέλη του ΤΙΚΑΦ πρόσφατα έρθαν και στην Επιτροπή σας και ανέφεραν τα σχετικά. Τώρα, Δεν θέλω να μπω σε άλλες λεπτομέρειες, αλλά να απαντήσω σε συγκεκριμένες σας απορίες. Να σας μιλήσω όμως για την ε, Αφρική και ιδίως τη Δυτική Αφρική, όπου έχουμε ισχυρή παρουσία, πιστεύουμε ότι για τα θέματα φύλου και SSR είμαστε από τους ε, πρωτοπόρους εκεί. Πραγματικά Είμαστε πάρα πολύ δεσμευμένοι και υπέρ του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Προσπαθούμε να δώσουμε στις κυβερνήσεις ε, οποιαδήποτε βοήθεια, εγχειρίδια, μελέτες και άλλα έγγραφα μπορούν να βοηθήσουν. Και είχαμε πρόσφατα δημοσίευσει την ε, ε, μελέτη για την κοινοβουλευτική εποπτεία. Έχουμε συνεργαστεί με κοινοβουλευτική συνέλευση της ΟΑΣΕ, IPU και άλλους. Θα συνεχίσω τώρα στα γαλλικά. Θέλουμε τώρα να συνεχίσουμε τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαιτέρως και μάλιστα με την δικιά σας υποεπιτροπή. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει, αλλά για μας θα ήταν μία μεγάλη χαρά να μπορέσουμε να υποδεχθούμε αυτή την υποεπιτροπή με μία εκδρομή που θα κάνετε στη Γενέβη για να μπορέσω να σας δείξω το τι κάνουμε, το κέντρο και τους συνεργάτες μας και ελπίζω ότι θα είναι κάτι που θα σας ενδιαφέρουν. Σας ευχαριστώ για ερωτήσεις και για παρατηρήσεις και κλείνω με αυτά τα σχόλιά μου. Ευχαριστώ κύριε ε, πρέσβη για τα σχόλιά σας διότι αυτά είναι πολύ χρήσιμα για πολλά από μας ε, χρησιμοποιείτε την πείρα σας και ε, πολύ όντως επηρεάζονται από τις γνώσεις σας και την εμπειρία του κλιμακίου σας. Έχω να κάνω δύο ερωτήσεις. Ε, θα ήθελα δηλαδή να ξέρω ποιο είναι το πρόγραμμά σας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο γιατί στην Επιτροπή αυτή ε, προσπαθήσαμε να υιοθετήσουμε μία συμφωνία σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που είναι ένα βασικό θέμα για την Επιτροπή μας και από την άλλη πλευρά ε, θέλω να αναφερθώ στην δημοκρατική εποπτεία διότι συζητήσαμε για τις συμφωνίες για τα PNR με τις Ηνωμένε Πολιτείε που είναι ε, μια συμφωνία πολύ λεπτή και ευαίσθητη αλλά ε, υπάρχει δυσκολία για δημοκρατική εποπτεία του Κοινοβουλίου Ποια είναι η δικιά σας γνώμη, γιατί πολλές ε, από τις δραστηριότητες γίνονται πιο διεθνείς, ε, πιο παγκοσμιοποιημένες και η κλασική εποπτεία δεν θα είναι τόσο αποτελεσματική. Ο κύριος Πάσκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, ε, δεν έχω τόσες ερωτήσεις γιατί εφόσον είμαι στη συμβουλευτική, ε, ε, στη συμβουλευτική επιτροπή που επιβλέπει το Συμβούλιο της ΔΙΚΑΦ παρακολουθώ. Αλλά χαίρομαι που ήρθε ο ο κύριος ε, μόνο και μόνο για αυτήν την ε, ε, συνάντηση ο πρέσβης κύριος Βίνκλερ διευθυντής της ΔΙΚΑΦ αλλά υπάρχει μια θεωρία από ό,τι ξέρω και ουσιαστικά χρειάστηκε όπως λέμε στο κασίδι το κεφάλι να μάθουμε από τα λάθη μας και να καταρτήσουμε ορισμένες αρχές διότι ε, ιδίως όσον αφορά το δημοκρατικό έλεγχο των στρατιωτικών δυνάμεων που είναι μία πρόκληση για την δημοκρασία γενικώ. Και μετά η Επιτροπή που ξεκίνησε το 2000 άρχισε να εργάζεται στενά με τις χώρες της κεντρικής ε, ε, Ευρώπης και σιγά σιγά άρχισε να κινείται προς τα Βαλκάνια και μετά ε, δραστηριοποιήθηκε εκτός Ευρώπης σε σημαντικά σημεία. Πρέπει λοιπόν να πω ότι με αυτόν τον τρόπο το Ινστιτούτο μπόρεσε αφενός να αποκτήσει αυτή την πρακτική εμπειρία και Βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και από την άλλη πλευρά ε, προσπαθεί να καταρτήσει ε, τις ε, ένα σύστημα από όλες αυτές τις πληροφορίες τις οποίες έχει συγκεντρώσει. Αντιλαμβάνομαι ε, άλλωστε εφόσον έχω συμμετάσχει στις αποστολές στην Ινδονησία, στην Καμπότζη και στην Ταϊλάνδη και σε άλλες, θα ήθελα να ξέρω πόσο ενδιαφέρον ε, υπάρχει σε αυτές τις χώρες για τέτοια μέτρα. Επίσης ε, το Ινστιτούτο ενδιαφέρεται επίσης και για τις καταστάσεις μετά από τις διαμάχες. Χαίρομαι που αποκαταστήσατε τις σχέσεις σας με την Τινησία. Διότι ήταν πολύ σημαντική η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να διαμορφωθεί οι δυνάμεις ασφαλείας, ιδίως σε χώρες αυτού του τύπου. Και αντιλαμβάνομαι ότι πριν από λίγους μήνες Είδαμε τον Hans Born, ο οποίος ε, ήρθε στο Κοινοβούλιο και παρουσίασε μία σημαντική θέση ε, σχετικά με τον τομέα ε, της, ε, των υπηρεσιών ε, ασφαλείας στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δηλαδή ε, διάφορα στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τις σχέσεις των διαφόρων Ινστιτούτων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι ότι αυτό το Ινστιτούτο το οποίο είναι ελβετική επιχείρηση είναι αδέκαστο και πολύ αντικειμενικό. Ευχαριστώ. Η κυρία Κοπά. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Κοπά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρέσβη για τη συνεισφορά σας. Ο δημοκρατικός έλεγχος των ενόπλων δυνάμεων είναι κάτι το πάρα πολύ χρήσιμο. Βλέπω ότι η Λευκορωσία εισήλθε το 2002. Εσείς πώς προωθείτε τα αποτελέσματά σας σε χώρες μέλη στις οποίες υπάρχουν προβλήματα σε επίπεδο κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ισορροπία. Πώς ακριβώς τα καταφέρνετε, Κρόνμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρον το κέντρο σας. Νομίζω ότι ο δημοκρατικός έλεγχος των ενόπλων δυνάμεων είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Αλλά τι γίνεται με το δημοκρατικό έλεγχο των ιδιωτικών στρατών και των ιδιωτικών εταιριών παροχής ασφαλείας. Νομίζω ότι είναι διπλή η δουλειά. Πώς θα ελέγξουμε αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες και από την άλλη ποιο είναι το καθεστώς του προσωπικού που εργάζεται στις εταιρείες αυτές. και που πρέπει να ελέγχονται από το διεθνές δίκαιο. Πώς βλέπετε εσείς το θέμα αυτό και τι μπορεί να γίνει. Πιστεύετε ότι η ευρωπαϊκή θέση πρέπει να αναλάβει κάποια δράση, ή τι πρέπει να κάνουμε σε σχέση με αυτές τις εταιρείε. Υπάρχει ανάγκη για διεθνείς συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για καθορισμό κριτηρίων σχετικά με τις δραστηριότητες των εταιριών. Δύο ερωτήσεις ακόμα. Ευχαριστώ για την παρουσία του τον κύριο Βίνκλα. Ελπίζω αυτό να ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα στο κοινοβούλιο μας και την ΤΙΚΑ. Γιατί εκτιμώ ιδιαίτερως τη δράση του Ινστιτούτου. Να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπε μόλις τώρα η κυρία Κρόνμπεργκ. Έγινε μια πολύ σημαντική έκθεση της ΔΙΚΑΦ υπογραμμίζοντας την πραγματικότητα αλλά και τους συνδύνους που ενέχει το θέμα της ε, συνεχούς διεύρυνσης του ρόλου των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής ε, ασφαλείας, υπηρεσιών ασφαλείας. Αυτή αυτό το outsourcing ουσιαστικά η, ε, θα έλεγα η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον τομέα της παροχής μέτρων ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σε δύο ώρες εγώ θα φύγω για να πάω στη Λιβύη με την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου και εκεί βλέπουμε όλα αυτά τα κοράκια θα έλεγα γύρω μας και διαρωτώ με λοιπόν τι γίνεται με την κατάσταση αυτή και ποια είναι η πραγματικότητα η οποία δικαιολογεί τη χρήση τέτοιου είδους ε, δυνάμεων. Εξετίμησα επίσης και την προσπάθεια την οποία έχετε κάνει για το δημοκρατικό έλεγχο. Αλλά δεν έχει υπάρξει δυστυχώς πρόοδος ούτε σε επίπεδο κρατών μελών, ούτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. και φυσικά εκεί που είχαμε συγκεκριμένο πρόβλημα ήταν με τις ε, μετακινήσεις κρατουμένων παρανόμους όπου, ανάμεσα στις χώρες της Ένωσης όπου δυστυχώς τίποτα δεν έγινε σοβαρά εκτός από την έκθεση την οποία είχε κάνει το ίδιο το Κοινοβούλιο. Που παρουσίαζε βέβαια και αρκετές αδυναμίες. σχετικά με τον ρόλο των γυναικών για την εφαρμογή της απόφασης των Ηνωμένων Εθνών Το θέμα της ισορροπίας των φύλων είναι ένα σημαντικό θέμα και στον τομέα των ενόπλων δυνάμεων. Ελπίζω να ξεκινήσει μια αξιολόγηση των ρυθμίσεων των νομοθετικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον έλεγχο της εξαγωγής οπλικών συστημάτων. Στάσκη, στάσνη, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Βίνκλερ, πρέσβη Βίνκλερ, για την παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες, ευχαριστούμε και την ελβετική κυβέρνηση, η οποία καλύπτει το 50% του προϋπολογισμού σας. Ίσως ιδιωτικές εταιρείες παρέχουν το υπόλοιπο. Ελπίζω να έχετε περισσότερα μέλη στην οργάνωσή σας και από τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό θα ήταν πολύ θετικό. Ε, είδα και τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις σας Κάποιες από τις εγκαταστάσεις είναι μόνιμες, κάποιες είναι προσωρινές, ιδιαίτερα στη Βηρητό. Αν παραμείνετε ας πούμε στη Βηρητό ή μάλλον ε, σκοπεύετε να παραμείνετε, πιστεύετε ότι έχει σημασία η παρουσία σας εκεί. ή πιστεύετε ότι θα πρέπει να πάτε καλύτερα σε χώρες όπου υπήρχαν παλιότερα αυταρχικά καθεστώτα όπως στη Βαγδάτη, στην Τρίπολη κτλ. Κύριε Δίνκλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, συγγνώμη. Θα απαντήσω μία προς μία και θα είμαι όσο μπορώ περισσότερο σύντομο. για την προοπτική μέχρι το 2015. εμεί στα πλαίσια του εγγράφου μας του στρατηγικού πέρυσι προσπαθήσαμε να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε, τι έχουμε μπροστά μας, ποια είναι τα χαρτιά που έχουμε μπροστά μας. Φυσικά δεν μπορούμε να προβλέψουμε το τι θα γίνει το 2015 αλλά για το 2000 ε, ή μάλλον το 2050 δεν μπορούμε να προβλέψουμε, αλλά το 2015 μπορούμε να κάνουμε κάποιες προβλέψεις. Έχουμε κάνει κάποιες μελέτες λοιπόν. Έχουμε λάβει υπόψη μας ε, διάφορα χαρακτηριστικά όπως οι, δημοκρατικές, οι δημογραφικές αλλαγές, Έχουμε επίσης σταθεί στο θέμα της συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε πολλούς τομείς και στον τομέα της ασφαλείας και στον τομέα του κυβερνοχώρου. Είναι περίπλοκο το θέμα Υπάρχει το μπίρχερ μουσλι που τρώμε στην Ελβετία στο πρωινό με γιαούρτι και φρούτα. Τα ανακατεύουμε και είναι συνηθισμένο πρωινό. Έχω τη συζήτηση λοιπόν ότι έχω την αίσθηση ότι η συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από τέτοια θέματα είναι ένα θέμα μείγματος αμαλγάματος πολλών διαφορετικών προβλημάτων. Δηλαδή ο κυβερνοπόλεμος είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί κατά καιρούς. Όσο πιο αναπτυγμένη είναι μια κοινωνία σε επίπεδο κυβερνοχώρου, τόσο πιο ευάλωτη είναι η κοινωνία αυτή. Και δεν ξέρω ακριβώς τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε στον τομέα αυτό. Υπάρχει επίσης η εγκληματικότητα λέει ο μιλητής. Καταλήγουμε να πούμε ότι δεν υπάρχει έλεγχος ουσιαστικά γύρω από τα θέματα αυτά. Είναι όμως μια κατάσταση αυτή η οποία επικρατεί στο θέμα της χρήσης του κυβερνοχώρου για εγκληματικές δραστηριότητες, η οποία προκαλεί σύγχυση. Τα κοινοβούλια ασχολούνται, αλλά τελικά ποιοι ασχολούνται πιο συγκεκριμένα, οι ένοπλες δυνάμεις, οι υπηρεσίες ε, ας πούμε ασφαλείας των ενόπλων δυνάμεων. υπάρχουν προβλήματα χρήσης ε, του κυβερνοχώρου για εγκληματικές όπως είπα δραστηριότητες ε, είτε σε επίπεδο πνευματικής ιδιοκτησίας είτε σε επίπεδο παραβίασης κωδικών ε, χρήσης πιστοτικών καρτών. Γι' αυτό λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές σε σχέση με το ποιος τελικά είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο του κυβέρνοχώρου και γενικότερα για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων στον συγκεκριμένο χώρο. Εδώ υπάρχει χώρος για κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ξέρετε ότι η Σύμβαση της Βουδαπέστης του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι το βασικό όπλο, θα πρέπει να ενισχυθεί και σε επίπεδο γεωγραφικής εφαρμογής και σε επίπεδο ε, διεθνούς συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά μπορεί να κάνει εδώ. Υπάρχει μια τρίτη διάσταση αρκετά πιο περίπλοκη. Είναι οι νέες δυνατότητες ε, που δίδει ο κυβερνοχώρος στην κοινωνία των πολιτών. Ε, σκεφτείτε σαν παράδειγμα τις φωτογραφίες οι οποίες ε, κυκλοφορούν από την Κόμσο όπου δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι ή την ενημέρωση από την πλατεία Ταχρήρ. Έχουμε να κάνουμε μια νέα πραγματικότητα σε σχέση με τη χρήση του κυβερνοχώρου. Και δεν έχουμε δομές για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα. Έχουμε ένα μεγάλο, θα έλεγα, εργοτάξιο εδώ, ελέγχου του τομέα ασφαλεία της χρήσης, της χρήσης του κυβερνοχώρου. Ο δημοκρατικός έλεγχος, και έρχομαι σε αυτό που είπατε κυρία Πρόεδρε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε γρήγορα. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος ο κοινοβουλευτικός έλεγχος σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Είμαστε όλο και περισσότερο συνδεδεμένοι και προσπαθούμε να ελέγξουμε τις αλλαγές αυτές, να δούμε πώς προχωράει η πραγματικότητα. Θα πρέπει τα κοινοβουλευτικά σώματα να προσπαθήσουν να συζητήσουν το θέμα του κυβερνοχώρου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αυτή τη φάση έχουμε δύο εντολές. Καταρχάς είμαστε, οι, θα έλεγα, αυτοί οι οποίοι προτείνουμε τρόπους εφαρμογής της σύμβασης του ΜΟΤΡΕ. 38 χώρες, αν δεν κάνω λάθος, συμμετέχουν, έχουν υπογράψει τη σύμβαση του ΜΟΤΡΕ λέγοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες για τη χρήση ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας και στη διαδικασία αυτή ελέγχονται οι σωστές πρακτικές οι οποίες θα πρέπει να γίνονται σεβαστές. Το κείμενο του Μοντρέ λοιπόν. Υπάρχει μια σχολή σκέψης η οποία λέγει και συμφωνώ με αυτήν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διεθνή σύμβαση που να υπογραφεί από όλε τις χώρες. Είναι μια καλή ιδέα, αλλά εκεί έχουμε μείνει. Είναι μια ιδέα, είναι θα έλεγα μια επιθυμία και υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες δεν επιθυμούν να υπογράψουν μια τέτοια σύμβαση. Δεν έχει ας πούμε υπογραφεί η συμφωνία του Μοντρέ, η σύμβαση μάλλον του Μοντρέ από την Αμερικανική κυβέρνηση. Εμείς ε, στην διαμόρφωση των διαπραγματεύσεων για τους συγκεκριμένους αυτές, ε, αυτούς, ε, αυτές ρυθμίσεις συμμετέχουμε. Υπάρχουν λίγες χώρες, λίγες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάντως προσυπογράψει τον σεβασμό, την δήλωση σεβασμού του συγκεκριμένου αυτού κώδικα συμπεριφοράς που προβλέπεται στη σύμβαση του ΜΟΤΕ. Εμείς προσπαθούμε σε αυτή τη φάση να δημιουργήσουμε έναν εφαρμοστικό μηχανισμό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κάποιες επιχειρήσεις που μετέχουν στον τομέα αυτό, που εμπλέκονται στον τομέα αυτό να προσυπογράψουν τον κώδικα, αλλά από την άλλη θα πρέπει να ελεγχθούν όλας για τον τρόπο σεβασμού των ρυθμίσεων που, που περιλαμβάνει ο κώδικας αυτός. Υποτίθεται ότι έχετε αναλάβει το σεβασμό σαν παράδειγμα της ε, σύμβασης της Γενέβης, ε, αλλά από την άλλη δεν έχετε σεβαστεί ακριβώς τις ρυθμίσεις, από ό,τι φαίνεται σε κάποιες από τις επιχειρήσεις σας, θα μπορούσαμε να πούμε στις ιδιωτικές εταιρείε. Απαιτείται λοιπόν ένας εφαρμοστικός μηχανισμός. Αυτή είναι η διαδικασία την οποία προσπαθούμε να προωθήσουμε. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Υπάρχει, ξέρετε, και η διαδικασία ελέγχου των δραστηριοτήτων ε, και του κώδικα συμπεριφοράς που πρέπει να σέβονται οι εξορικτικές επιχειρήσεις, οι εξορικτικές δραστηριότητες συμμετέχουμε στην προσπάθεια επεξεργασίας ενός ε, κειμένου σχετικά δεσμευτικού. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε τις προθέσεις αυτών που θέλουν ε, μια ευρύτερη διεθνή σύμβαση για τη χρήση των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας πάντως. και δημιουργούμε πρότυπα νομικών ρυθμίσεων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Τα κείμενα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν και να γίνουν δεκτά όχι μόνο σε αυστηρά νομοθετικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο πολιτικό βέβαια. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Ιων Πάσκου για τα καλά του λόγια. Βλέπω εδώ και άλλους παλιούς φίλους. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε την ε, ταπεινή μου παρουσίαση. Να πω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην αγνοούμε κάποιες διαστάσεις. συνολικά Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων στον τομέα ασφαλείας. Όχι μόνο ένοπλες δυνάμεις, αλλά και ιδιωτικές φυσικά επιχειρήσεις. Να παρακολουθούμε περιπτώσεις μετάβασης προς τη δημοκρατία με τα συγκρουσιακές καταστάσεις που διαμορφώνονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, παρακολούθηση των δραστηριοτήτων στον κυβέρνοχώρο, η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σύνθετη και θα πρέπει να μην την αγνοούμε. Ώσπου να τελειώσει ένα σεμινάριο πάνω σε ένα α θέμα έχει ανοίξει ένα β. Θέλουμε λοιπόν εμείς αυτά τα πακέτα συζήτησης τα οποία έχουμε διαμορφώσει να αποκτήσουν μια κάποια χρονική διάρκεια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πραγματικότητας. Έτσι ερχόμαστε και στον ορίζοντα του 2015 σε σχέση με τις διεθνείς συμβάσεις, σε σχέση με τις συζητήσεις για τον έλεγχο στον κυβέρνο χώρο. Απαιτείται συντονισμός καλύτερο σε επίπεδο εντοπισμού των βέλτιστων πρακτικών συντονισμού των διαφόρων εμπλεκομένων Ελπίζω ότι η δομή μας σαν ίδρυμα να μπορεί να συνδυάσει την δυνατότητα που έχει μία μη κυβερνητική οργάνωση που είναι ευαίσθητη και ευέλικτη στην ανταπόκριση στις, δημιουργούμενες καταστάσεις, από την άλλη όμως να έχουμε και τη σταθερότητα και τη διάρκεια που απαιτείται για να μην λειτουργούμε αποσπασματικά. Η πρόκληση λοιπόν είναι μεγάλη. Πολλά εργοτάξια είναι μπροστά μας και η ζήτηση για τις υπηρεσίες μας αυξάνεται με εκρηκτικό ρυθμό και αυτό μας επιβαρύνει αλλά κυρίως μας δίνει πάρα πολλές ευθύνες. Υπάρχουν δύσκολες περιπτώσεις όπως η Λευκορωσία. Πώς να ασχοληθεί κανείς με την περίπτωση της Λευκορωσίας. Ζήτησε να γίνει μέλος και του δώσαμε τη δυνατότητα αυτή με στόχο να αποκαταστήσουμε γέφυρες με τη λευκορωσική πραγματικότητα. Οργανώσαμε παρόλα αυτά κάποιες, κάποια σεμινάρια στο Μίνσκ, αλλά δεν έχουμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχουν πετύχει τους στόχους μας. Αλλά παρόλα αυτά βαραίνουμε στην κατάσταση όσο μπορούμε και ελπίζουμε να μπορέσουμε να επηρεάσουμε κάποιες αλλαγές προς σωστή κατεύθυνση. για τα σχόλια της κυρίας Γκομές σχετικά με τη χρήση των ιδιωτικών υπηρεσιών. Προφανώς υπάρχει πίεση προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι σαφές ότι οι ιδιωτικές ε, επιχειρήσεις ασφαλείας αυξάνονται συνεχώς και αναπτύσσονται συνεχώς. μειώνεται ο αριθμός των στρατευμάτων σαν παράδειγμα σε περιπτώσεις επέμβασης όπως το Αφγανιστάν, αυτό θα αυξήσει τις ιδιωτικές εταιρείες, την προσφυγή στις υπηρεσίες τους. Γενικά οι επιχειρήσεις ασφαλείας συνεργάζονται στις προσπάθειες διαμόρφωση αυτού του κώδικα οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξουν καθορισμένες ε, πρακτικές. Αλλά απαιτείται πάρα πολύ δουλειά. Τα SSR και SSG. Εδώ νομίζω ότι η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφής. Εμείς φυσικά προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να αναλάβει δράση. Ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο σχεδιασμού των δράσεων και σε επίπεδο πρακτικό θέτουμε στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα μέσα τα οποία έχουμε τα αναλυτικά εννοώ, αλλά απαιτείται μια επεξεργαστική δράση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που για μας είναι και παραμένει θα έλεγα βασικός εταίρος. θα είμαστε στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα τα προγράμματα με τα οποία ασχολείστε. Για τις εγκαταστάσεις μας. Έχουμε, γραφεία και εδώ στις Βρυξέλλες. Έχουμε επίσης γραφεία στη Λιουμπλιάνα. Στις Βρυξέλλες έχουμε ένα άτομο. Και είναι κοντά στις Γενέβη και αν χρειάζονται εμπειρογνώμονες έρχονται εδώ αλλά έχει τοπική νομική υπόσταση το γραφείο μας αυτό. Στη Λιουμπλιάν έχουμε το γραφείο που παρακολουθεί τη δράση των αστυνομικών δυνάμεων. Συνεργαζόμαστε με εμπειρογνώμονες αστυνομικούς από τη Σερβία, τη Βοσνία. Στη Βηρητό είναι μια αποστολή η οποία δεν έχει, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη νομική ταυτότητα και δεν υπάρχει συμφωνία από πλευράς, της, ε, πλευράς του Λιβάνου για το πώς θα προχωρήσουμε σχετικά με την αναγνώριση, θα έλεγα, αυτής της ε, αποστολής της υπηρεσίας. Ραμάλα, 14 άτομα, μεγάλη παρέμβαση και στη Λουμπλιάνα έχουμε γύρω στους 12. Είμαστε σε στενή συνεργασία και με τις ε, δυνάμεις των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ραμάλα, με τους εκπροσώπους μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ραμάλα. Υπάρχει θέμα με το κράτος δικαίου και τη σωστή λειτουργία των συνθήκων ασφαλείας στην Παλαιστινιακή πραγματικότητα. Είναι πολύ περίπλοκη η Παλαιστινιακή πραγματικότητα. Την είδα έξι άτομα, θα φτάσουν τους 12 όπου να είναι στο γραφείο μας. διαπραγματευόμεθα σε αυτή τη φάση όλους τους εμπλεκομένους, με όλους τους εμπλεκομένους και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την κυβέρνηση Άλλωστε έχω και το απόγευμα επαφές με την Κομισιόν. έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κάτι που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Τινησίας. Έχουμε επίσης και ένα μικρό γραφείο στην Αμπούζα, που ασχολείται με τα θέματα της Δυτικής Αφρικής. Τώρα για την περίπτωση δημιουργίας τέτοιου είδους ε, εγκαταστάσεων στην Τρίπολη ή αλλού. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε αρκετά ευέλικτοι. Μπορεί να ανοίξουμε γραφεία, μπορεί να κλείσουμε κάποια αν δεν είναι πλέον χρήσιμα. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι η Τίνιδα ίσως θα μπορούσε να εξυπηρετήσει την περιοχή να είναι ένα κέντρο συντονισμού δραστηριοτήτων. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα προχωρήσουμε, τι θα γίνει, αν θα πρέπει να πάμε κάποια στιγμή στο Μαρόκο ή στη Λιβύη. Θα πρέπει να λάβουμε πάρα πολλά πράγματα υπόψη μας ε, πριν ε, ανοίξουμε κάποιο γραφείο. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και η αποστολή στη Λιβύη την επόμενη εβδομάδα ίσως μας διαφωτίσει περισσότερο. Υπάρχουν άλλα ερωτήματα αγαπητοί συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω τότε τον πρέσβη. Νομίζω ότι η σημερινή μας συνάντηση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είχαμε μια πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Όπως προείπα, το κέντρο δημοκρατικού ελέγχου των ανόπλων δυνάμεων είναι πολύ κοντά σε εμά. Χαιρόμαστε λοιπόν όποτε προσφεύγουμε και χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες σας. Η ανταλλαγή καλών πρακτικών φυσικά ε, είναι πολύ σημαντική και εσείς μας βοηθάτε να γνωρίζουμε τις καλές πρακτικές, να μπορούμε και να τις ανταλλάσσουμε βέβαια. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και για την πρόσκληση. Η Επιτροπή μας φυσικά ε, και ενδιαφέρεται να μεταβεί στη Γενέβη για να μπορέσουμε εκεί να έχουμε μια ακόμη πιο ευρία ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Thank Colleagues, the next point αγαπητοί συνάδελφοι, επόμενο με τη μερισιά διάταξη είναι η αντιπροσωπεία τη Επιτροπή ε, ΣΕΝΤΕ στη Βαρσοβία. Ξέρετε ότι στι 15 και 16 Δεκεμβρίου είχαμε μια αντιπροσωπεία εκεί, στην Βαρσοβία. Πρασάτζιτ και Γιάννη ήταν στη Βαρσοβία εκ μέρου τη Επιτροπή μα. Η γραμματεία έχει ήδη εκπονήσει την έκθεση δεν ξέρω αν θέλουν οι συνάδελφοι να αναφέρουν κάποια πράγματα. Κύριε Γιάννης, αν θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ουσιαστικά απλά από ευγένεια ε, παίρνω το λόγο γιατί η έκθεση που έχουμε στο φάκελό μας και την οποία εκπώνησε η γραμματεία είναι πάρα πολύ αναλυτική. Ήμουν ο στην ε, συνάντηση αυτή. Μαζί με την κυρία Γησάγκη πήγαμε στις 15 και 16 η Μπρισάτζιτς. Λοιπόν, πήγαμε με την κυρία Μπρισάτζιτς στην ε, Βαρσοβία 15 και 16 Δεκεμβρίου. Στόχος αυτού του ταξιδιού ήταν να δείξουμε στο τέλος της Πολωνικής Προεδρίας την αναγνώρισή μας από την πλευρά της Υποεπιτροπής μας ε, για το έργο, για την ηγεσία που επέδειξε η Πολωνία στα θέματα που μας απασχολούν, στα θέματα της πολιτικής ε, άμυνας, ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής. Το είπαμε λοιπόν, επισκεφθήκαμε το Υπουργείο Άμυνας, το Κοινοβούλιο και το ΓΕΘΑ της ε, χώρας, στη Βαρσοβία Μιλήσαμε και για την πρωτοβουλία της Βεϊμάρης που ανέλαβε η Πολωνία. Ήδη αριθμεί πέντε χώρες η πρωτοβουλία. Αριθμούσε τότε Γερμανία, ε, η Πολωνία και η Γαλλία ήταν οι ιδρυτικές χώρες. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι επειδή σας μιλάει ένας πολύ ένθερμος υποστηρικτής της κοινοτικοποίησης της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, πρέπει να σας πω ότι με πολύ μεγάλη χαρά βρήκαμε συνομιλητές σε αυτή τη πολύ μεγάλη χώρα, ε, την Πολωνία, που ήδη ε, ασκούν αυτή την πολιτική. Βέβαια, ε, ξέρουμε ότι ούτε και οι 27 χώρες, ούτε και όλοι οι τομείς είναι προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά βλέπουμε ότι όλο και μεγαλύτερη είναι η κρίσιμη μάζα που εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν λοιπόν βιώνουμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης και ξέρουμε πόσο ε, πρόβλημα υπάρχει ε, με τον αμυντικό προϋπολογισμό, που όχι απλά δεν μπορούμε να τον αυξήσουμε αλλά χρειάζεται και να περισταλεί σε πολλές ε, περιπτώσεις. Πρέπει λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την συγκυρία να μειώσουμε αλλά να μπορέσουμε και να, να συναθρήσουμε κατά κάποιο τρόπο, να συγκεντρώσουμε τις ε, δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε. Να έχουμε δηλαδή μια βέλτιστη χρήση των ε, πενιχρών μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Θέλουμε λοιπόν να, ε, πούμε ότι ήταν πάρα πολύ θετικά τα αποτελέσματα της σύντομης αυτής επίσκεψης. Σας ε, μετέφερα το περιεχόμενο, αλλά μπορείτε να το διαβάσετε και στην έκθεση που έχει διανεμηθεί ζούλευτες. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και σένα για την, αυτή την παρουσίαση. Λοιπόν, θα ξανασυνεδριάσουμε στις 28 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα στην ημερησία διάταξη, επομένως μπορούμε να κλείσουμε τη συνεδρία. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.